Por favor, tomen asiento, que vamos a continuar la reunión. El punto, el punto siguiente es la gestión actual y futura de la pesca en el Mar Negro, del que es ponente la señora Yotova. Ah, sí, la pesca, sí, la sé, perdón. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Σημείο 11. Καταπολέμηση παράνομη αλληλεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ρόλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκήτρια κυρία Λέβιν. έχουμε ένα έγγραφο εργασίας εκ μέρους της το οποίο θα μας παρουσιάσει. Thank you very thank you for everyone. Ευχαριστώ. πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Είναι ένα πρώτο έγγραφο εργασίας από τα δύο που θα έχουμε. Το συγκεκριμένο έγγραφο εργασίας εξετάζει την παρούσα λειτουργία των πόδα και τα μέτρα εναντί της ε, αλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι ιδιαίτερα επίκαιρο όταν μιλάμε για την πάταξη της παράνομης λαθρέας ε, αλίας ε, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βάση ε, από την οποία ξεκινούμε όταν ε, αντιμετωπίζουμε την πλάση παγκόσμιο επίπεδο είναι η πόδα. Είναι οι μόνοι οργανισμοί, οι μόνες οργανώσεις ε, που στα διεθνή υδατά στην ανοιχτή θάλασσα έχουν την αρμοδιότητα. Πόσες πόδα υπάρχουν για να σας πω πώς έχουν τα πράγματα. Είναι 18 αυτή τη στιγμή, 5 έχουμε εξετάσει καλύτερα και εξετάζουμε συγκεκριμένα ποια είναι τα μέτρα που χρησιμοποιούν για την παρά... πάταξη της παράνομης λαθρέας άναρχης αλίας. Αν έχετε το έγγραφο, μπορείτε να πάτε στην σελίδα 3. Ελπίζω να το έχετε το έγγραφο έγχρωμο. Υπάρχουν ε, κάποιοι χάρτες που δείχνουν ε, τον κόσμο και πάνω βλέπετε την κάλυψη των πόδων για τον τόνο και τα τονοειδή. Είναι μια εκπληκτική κάλυψη, σχεδόν όλο τον κόσμο καλύπτει και πρόκειται μόνο για το τονοειδή. Κάτω βλέπουμε την κάλυψη άλλων πόδα για άλλα αποθέματα και δεν είναι όλα που εμπίπτουν στην σύμβαση και όλες ε, οι ε, ελαφρώς γκρίζες εποχές ε, ρυθμίζονται εκτός από τις οικονομικές ζώνες των χωρών. Στη σελίδα 2 ναι, έχετε εκεί την ε, τρέχουσα έκδοση. Έχουμε κόκκινες περιοχές ε, που είναι η θάλασσα στον κόσμο που δεν εμπίπτει στους ρυθμιζόμενες περιοχές των πόδα Δηλαδή μπορεί κανείς να τις εκμεταλλευτεί, δεν υπάρχει ρύθμιση, δεν υπάρχει ελάχιστη προστασία. Τι κάνει μια πόδα όταν ε, πρέπει να πατάξει την παράνομη λαθρέα αναρκελία. Εξετάσαμε την ICAT που τη γνωρίζετε όλοι για τον ερθρό τόνο και άλλα τον ΟΕΔΗ. Από το 79 υπάρχει συγκεκριμένη ε, πόδα. Επίσης εξετάσαμε την, ε, το Οργανισμό Αλίας Νοτιοδυτικού Ατλαντικού, ε, την Επιτροπή Αλίας Δυτικού Κεντρικού Ειρηνικού μάλλον, την ΕΑΦΚΑ, την ΕΙΦΟ που έχουν μόνο βιομηχανικά κράτη και την ΚΑΜΛΕΡ, την Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θαλασσίων Αβιών Πόρων της Ανταρκτικής που έχουν ε, μεγάλη εμπειρία με τον τόνο της ε, Παταγωνίας και άλλα τέτοια ψάρια. Οπότε ποια είναι τα μέτρα που μπορούν να εφαρμόσουν οι υπόδερ. Αν δείτε το έγγραφο θα δείτε καταρχάς ε, την, τον εντοπισμό των πλοίων, κάτι που δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά και οι πέντε πόδα που είδαμε απαιτούν ε, να υπάρχουν ε, φάο ε, σημάνσεις, επισημάνσεις για τα πλοία που ελιεύουν εντός των υδάτων της δικαιοδοσίας τους. Επίσης υπάρχουν λίστες πλοίων που εξοδοτούνται να αλλιεύουν στην περιοχή που ρυθμίζει η πόδα και ονομάζονται άσπρες λίστες. Αν δεν είναι στη λίστα ένα ε, πλοίο που δράσει την περιοχή θεωρείται ότι είναι παράνομο. Όλες οι πόδα έχουν τέτοιες λίστες, αλλά είναι διαφορετικές. Η ICAT, ας πούμε, καλύπτει μόνο πλοία άνω των 20 μέτρων. Η WCPFC, η ΝΕΦΚΑ, η ICAT περιλαμβάνουν επίσης τα ψυγεία και τα φορτηγά, όχι όμως οι άλλοι. Και μετά έχουμε και τις μαύρες λίστες, που συμπληρώνουν τις άσπρες αλλιεύουν στην καλυπτόμενη περιοχή πλοία, δηλαδή χωρίς άδεια, τα οποία εικάζεται ότι προβαίνουν σε παράνομη λαθρέα αναρχή αλία. Υπάρχουν άλλα που έχουν εξουσιοδότηση αλλά αλλιεύουν παράνομα. Εμφανίζονται επίσης ε, τέτοια πλοία τα οποία δεν μπαίνουν στα λιμάνια γιατί δεν έχουν αυτή την άδεια και όλα τα μέτρα ενημερώνονται με πολύ αργό ρυθμό. Οι λίστες επικαιροποιούνται μόνο κατά την ετήσια συνάντηση και μπορεί να είναι πολύ πολιτική η κατάλογη. Ο καθένας προσπαθεί να κρατήσει τα πλοία του εκτός λίστα. Οπότε στη μαύρη λίστα είναι τα πλοία που δεν, είναι στα δεν ανήκουν στα συμβαλώμενα μέρη. Αυτή τη στιγμή η ICAT ε, απαριθμεί 24 πλοία, 21 αγνώστου σημαία, ένα από τη Γουινέα και δύο από τη Βολιβία. Ένα άλλο μέτρο που χρησιμοποιούν και οι πέντε πόδα που εξετάσαμε είναι οι εμπορικές κυρώσεις. Η ICAT κυρίω χρησιμοποίησε αυτό το μέτρο, το οποίο όμως τελικά φάνηκε ότι ήταν πολύ δύσκολο. Στη δεκαετία του 90 απαγόρευσε την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από τις χώρες εκείνες που οι σημαίες τους, τη έφεραν ε, σκάφη χωρίς εξουσιοδότηση. Από το 2008 χώρες ε, είχαν υποστεί αυτές τις απαγορεύσεις εισαγωγών. Όμως, βραχίδια τα αποτελέσματα γιατί τα πλοία μεταπίδησαν σε σημεία άλλων χωρών που δεν υφίστανται κυρώσεις. Οι χώρες που υφίστανται κυρώσεις τις αφαιρούσαν προσχωρώντας την ΕΚΑΤ. Έτσι λοιπόν, ε, είχαμε το επόμενο μέτρο, το να επιθεωρήσεις στη θάλασσα, όπου μόνο οι ναύκο και αυκά πετούν από τα συμβαλόμενα μέρη να αποστέλουν πλοία επιθεώρηση στη θάλασσα για την αλία στην οποία συμμετέχουν. Είναι δηλαδή ε, εθελούσε η συμμετοχή στις άλλες περιπτώσεις. Ε, τώρα, παρατηρητές πάνω στο πλοία. Μόνο η ΝΕΙΦΟ να ένα παρατηρητή ένα πλοίο. Η ΆΙΚΑΤ, μόνο για τα εχθειοτροφία ερθρού τόνου. Ε, για τα γρηγρή και για τα πλοία ψυγεία. Μέτρα κράτους λιμένα και αυτά σημαντικό εργαλείο έχουν συμφωνήσει η πόδα ότι κάθε κράτος θα πρέπει να προσέχει ποια είναι τα ψάρια που εκφορτώνονται στα λιμάνια τους η WCPFC δεν έχει βέβαια τέτοιες ε, απαιτήσει για επιθεωρήσεις στο λιμάνι, αφήνοντας το στη διακριτική ευκαιρία του κράτους λιμένα. Οι άλλες έχουν διαφορετικούς κανόνες. Συστήματα τεκμηρίωσης των αλλιευμάτων, η ICAT και η CAMLAR το έχουν, αλλά όχι οι υπόλοιπε. Ναύλωση πλοίου. μπορεί κανείς να αναβλώσει, ένα συμβαλόμενο μέρος να αναβλώσει ένα ε, πλοίο από μήνυ ε, συμβαλόμενο μέρος, ε, το οποίο δημιουργεί προβλήματα με τις ευθύνες του κράτους που ναυλώνει. ειδικότερα για χώρες που δεν έχουν θαλάσσια παράδοση. Μόνο η ICAT και η ΝΕΦΟ προσπάθησαν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Η, μεταμόρφωση, η μεταφόρτωση επίσης είναι κάτι που χρησιμοποιήθηκε. Ειδικότερα όταν όμως γίνεται στη θάλασσα υπάρχει ένα κενό ε, που επιτρέπει παράνομη λαθρέα αρναρχελία. Η ΆΙΚΑΤ έχει μια γενική απαγόρευση για τις μεταφορτώσεις στη θάλασσα, οι άλλες ε, ε πόδα όχι. Αυτά ήταν που εξετάσαμε για τη σπόδα. Τι βρήκαμε. Είδαμε ότι προχωρούν τα πράγματα, εξελίσσονται αλλά αργά και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι παρόλο που κάποια μέτρα έχουν υιοθετηθεί από τη σπόδα δεν τα εφαρμόζουν πάντα τα συμβαλόμενα μέρη. Εάν τα μέτρα αυτά δεν μεταφράζονται σε ε, εθνική νομοθεσία από τα συμβαλόμενα μέρη είναι δύσκολο κανείς να συμμορφωθεί όταν έχουμε ας πούμε ελέγχους ε, στους λιμένες ε, κτλ. Η αλλαγή λοιπόν είναι θέμα βασικά πολιτικής θέλησης και ένα κέριο πρόβλημα με τη σπόδα είναι η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν υπάρχουν δεσμευτικές υποχρεώσεις αυτή τη στιγμή ε, για την διατήρηση των βιολογικών έμβιων πόρων, δηλαδή στην στα ύδατά του. Σε κάποιες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία, αλλά ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις ε, βλέπουμε ότι γίνεται σπάνια, ε, συνήθως είναι η συνένεση και πάντοτε, ακόμα και στην πλειοψηφία, προσπαθούν να αποτρέψουν τον καθένα από τον ψηφίσει όπως ε, θέλει. Πώς θα αλλάξουμε την εικόνα λοιπόν. Αυτό που είναι κοινή ε, παγκόσμια κληρονομιά, ε, οι θαλάσσιοι πόροι δηλαδή, πώς μπορούν να προστατευτούν. Η πόδα θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογούνται τακτικά από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Οι αξιολογήσεις και όλα τα στοιχεία θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανή η εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται από τις αξιολογήσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τις εμπλεκόμενες πόδα ιδανικά και αυτό δεν το λέω σαν γραφεργασίας Η ιδέα ίσως ενός νέου ε, φορέα στο σύστημα του ΟΗΕ θα μπορούσε να δοκιμαστεί και να θεσπιστεί και ίσως αυτό το σύστημα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις ανεξάρτητες αυτές ε, επιθεωρήσεις των ε, πόδα για να υπάρχουν και εναρμονισμένα κριτήρια και στάνταρτ. Και όταν δεν συμμορφώνεται κανείς ε, να υπάρχουν κυρώσεις όπως μείωση ποσοστώσεων, εμπορικές κυρώσεις κτλ. Με αυτόν τον τρόπο το κάθε κράτος θα πιέζεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες. Πώς θα συμφωνήσουν ε, τα συμβαλώμενα μέρη, βέβαια τον πόδα, να εξετάζονται και να επιθεωρούνται. Θεωρώ ότι ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων ανήκουν σε πλά ε, αλία και αυτό είναι με μια μεγάλη κλοπή. Μιλάμε για φοροδιαφυγή, για διάφορα τέτοια προβλήματα, ε, για πλοία που έχουν σημαία μίας χώρας, ε, που ανήκουν σε offshore, σε φορολογικούς παραδείσους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά είναι παγκόσμια ζητήματα, ένα σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε διεθνές επίπεδο. Αυτοί που ουσιαστικά ασκούν την παράνομη αλληλεία δρούν σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά οι, όσοι τους ελέγχουν δεν το κάνουν. Πρέπει να θεωρηθεί και παγκόσμιο ευρωπαϊκό, ε, μάλλον συγγνώμη, παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα που ε, πλήττει το θαλάσσιο οικοσύστημα και η παγκόσμια κοινότητα θα μπορούσε και θα πρέπει να απαιτήσει να γίνεται διαχείριση αυτών των πόρων με ελεγχόμενο και βιώσιμο ε, τρόπο. Πρέπει να ανεχνεύονται τα ύποπτα ε, είδη και τα ύποπτα σκάφη και να υπάρχει και ένας παγκόσμιος κατάλογος το οποίο είναι κάτι που συζητείται, αλλά δεν έχει ακόμα αποφασιστεί. Θα αποφασιστεί από τον ΦΑΟ ίσως την επόμενη εβδομάδα. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός. Πρέπει να έχουμε ηγετικό ρόλο, γιατί είναι η μόνη αλληλευτική δύναμη που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. να εφαρμόσουμε τον νέο κανονισμό για την ΠΛΑ από όλα τα κράτη, να εφαρμόζεται ο κανονισμό από όλα τα κράτη-μέλη και να κοιτάξουμε τι γίνεται και στη δική μας αυλή πρώτα και μετά να προχωρήσουμε. Πρέπει να ρωτήσουμε την Κομισιόν ε, να μας πει ε, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει ενθουσιασμός από τα κράτη-μέλη ως προς την εφαρμογή γιατί και με τη σπόδα το ίδιο ισχύει. Ε, οι κανονισμοί είναι καλοί όσο εφαρμόζονται. Θέλουμε να έχουμε καλά παραδείγματα στις εγχώριες περιοχές και αυτό θα βοηθήσει να έχουμε αποτελέσματα γενικώ. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την ε, Ισαμπέλα Λεβίν για την ε, εξαίρετη εισαγωγή της πολύ καλό το έγγραφο εργασίας που μας υπέβαλε, όμως οι τελευταίες παρατηρήσεις που κάνατε πραγματικά ε, περιγράφουν σωστά το πρόβλημα. Πρόκειται για ένα εγκληματικό φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, πρόκειται για πειρατική αλία. Αυτοί οι άνθρωποι συχνότατα χρησιμοποιούν ε, απαρχαιωμένων ελευτικά σκάφη και αλλιεύουν για πολλούς μήνες το χρόνο με κίνητρο να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους ε, με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Με αυτό τον... Ε, ε, μάλιστα πολύ συχνά προσλαμβάνουν αλληλείς από την Δυτική Αφρική, από παράκτιες περιοχές με μισθούς προσφέρουν 200 δολάρια το μήνα για παράδειγμα ε, που για αυτούς ε, ε, είναι τεράστιο ποσό, τους βάζουν σε αυτά τα αλληλευτικά, επικίνδυνα και απειχιωμένα αλληλευτικά σκάφη και τους λένε ότι το κόστος για την διατροφή τους και <laughs> για τη φιλοξενία τους στο σκάφος είναι παραπάνω από 200 δολάρια το μήνα ε, οπότε τους χρωστάνε δίθεν κιόλα. Τους αφαιρούν τα διαβατήριά τους για τις ταυτότητές τους και ζουν σε άθλιες συνθήκες πάνω σε αυτά τα πλοία. Αυτά τα πλοία ε, δεν γυρίζουν στη στεριά για πολλούς μήνες ε, διαμετακομίζουν τα παράνομα λευματά τους σε ε, φορτηγά ή ψυγεία ε, δεν ελέγχονται από κανέναν κανένας δεν γνωρίζει τις συνθήκες εργασίας των πληρωμάτων η, το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης ανακάλυψε ένα πλοίο το οποίο έφερε 200 εργαζόμενους που ζούσαν σε κάτι ξύλινες ε, ε παραγκούλες ε, στο πίσω μέρος του πλοίου που ζούσαν εκεί σε άθλιες συνθήκες, ε, υγειονομικές και άλλες. Μάλιστα ε, υπάρχουν καταγγελίες ότι οποιοδήποτε προσπαθήσει να εγκαταλείψει το πλοίο ε, δολοφονείται και το πτώμα του πετάγεται στη θάλασσα ε, ή πρόκειται για έγκλημα. Ε, οι άνθρωποι αυτοί κλέβουν αλλιεύματα, χρησιμοποιούν απαγορευμένα, απαγορευμένες αλλιευτικές τεχνικές και εργαλεία, και τεχνικές οι οποίες ε, ταυτόχρονα έχουν παρεμπίπτοντα αλλιεύματα τεράστια, ε, σκοτώνουν ε, χελώνες, θαλάσσιες και πολλά άλλα προστατευόμενα είδη. Και όπως είπε η Ισαβέλα, χρησιμοποιούν σημαίες ευκαιρίες και θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί και ορισμένα ευρωπαϊκά πλοία φέρουν τέτοιου είδους σημαίες ευκαιρίες, γιατί η Κομισιόν θα πρέπει να γνωρίζει ποια, ποια είναι αυτά τα πλοία. Υπάρχουν κατάλογοι με αυτά τα πλοία γιατί χρησιμοποιούν σημαίες του Παναδά, Παναμά, της Ονδούρας και των Γρεναδίνων νήσων ε, ε, ε, ευρωπαϊκά αλευτικά σκάφη. Και ευρωπαϊκοί λιμένες όπως η, το αυτός του, της Λασπάλμας στη, στα Κανάρια νησιά χρησιμοποιούνται ως λιμένες ευκαιρίες, ευκαιρίας. Πολλοί πολλά από αυτά τα σκάφη των ε, πειρατικών ελευτικών στόλων ε, ε, έχουν ως έδρα την Λασπάλμας. Και πολλά από αυτά τα παράνομα αλλιεύματα αναμειγνύονται με νόμιμα αλλιεύματα, φτάνουν στους λιμένες μας και πολλούνται σε εμά οι οποίοι τα αγοράζουμε. Πολλοί από εμά αγοράζουμε αυτά τα παράνομα αλλιεύματα χωρίς να το ξέρουμε και βέβαια το όλο αυτό φαινόμενο δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα στους νόμιμους αλλοίς. Ε, ταυτόχρονα όμως αγοράζοντας αυτά τα αλλιεύματα τροφοδοτούμε όλα αυτά τα φαινόμενα καταπίεσης και αθλειότητας που συμβαίνουν με, τους, με τα πληρώματά τους. Δεν θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και αν... Ο, ε, Κανείς άλλος δεν ε, μπορεί να το πετύχει, εμείς μπορούμε να πιέσουμε. Το 80% των παγκόσμιων αλλιευμάτων ε, τη χάνουν πλήρω εκμετάλλευση ή υπερεκμετάλλευση. Το οποίο σημαίνει ότι αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο θα καταρρεύσουν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την Ισαμπέλα για την ποιότητα της δουλειάς της και της έρευνας που έκανε. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Το έγγραφο είναι πάρα πολύ καλά διαρθρωμένο. Αναρωτιέμαι σε μία πρώτη φάση αν υπάρχουν οι ΟΕΡΠΕ, οι οργανώσεις οι οποίες μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες ή κυβερνήσεις που έχουν στατιστικά στοιχεία. Πολλές φορές είναι δύσκολο να έχουμε στοιχεία διότι δεν έχουμε εμείς τα πλάνα ε, ε και δεν ξέρω μήπως θα έπρεπε να απαγορεύσουμε την εισαγωγή από χώρες ε, οι οποίες δεν έχουν τα μητρώα τους πλήρη και δεν κάνουν τίποτα για την προστασία των ηχθικών τους πόρων. Εγώ έχω κατά νου εδώ και μία χώρα που επισκεφθήκαμε πρόσφατα τη Μαυρικανία που είναι μία χώρα λα, ε, λα ε, ξέρουμε ότι μαζί με τη Γεμένη ευνοούν την ε, αλία των Κινέζων ξέρουμε πολύ καλά ήμασταν ξέρουμε πολύ καλά που πάει το κατεψυγμένο ψάρι ε, των ε, κινέζικων πλοίων έρχεται στην Λασπάλμας και μετά από εκεί πάει στην Ευρώπη αυτό είναι ένα παράδειγμα μεταξύ των άλλων και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα το Μαρόκο έχει βέβαια μια διαφορετική χρειά το πράγμα είναι λίγο διαφορετικό το πρόβλημα αλλά σήμερα Υπάρχει ένα πρόβλημα, ένα διατροχό... Α, όλα απεγκλωβίστηκαν. Απίθανα, απίθανα. Διότι άμα δεν ε, είχε ε, ξεμπλοκαριστεί ε, η συμφωνία, αυτό θα είχε ευνοήσει την αλία της Ιεμένης. Επίσης έχω κατά νου και την Παπουασία Νέα Γουινέα συζητήσαμε ε, εχθές για αυτήν η οποία εξάγει όσα και αλλά για τον τόνο και άλλα προϊόντα τα οποία κονσερβοποιούνται ε, δεν χρησιμοποιεί, δεν κάνει αυτή τη χρήση. Θα ήθελα λοιπόν να συνεννοηθούμε για αυτόν τον τομέα και με τις άλλες χώρες του ειρηνικού για την, παρέ, για την παρέκκληση στους κανόνες προέλευσης Δεν μιλάω εγώ για την υπόλοιπη συμφωνία η οποία είναι εντάξει αλλά για τον κανονισμό ελέγχου κατά της αλίας πλά Ο κύριος Αρσένης. And, uh, I would like to Ευχαριστώ θερμά την Ισαβέλα για αυτή τη, τη δουλειά. Με όλες αυτές τις ε, λεπτομέρειες ε, έχουμε μια πραγματικά πολύ καλή βάση για να συζητήσουμε αυτό το καινούριο θέμα για την Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε λοιπόν. Θα συμφωνούσα και με τον Στιόρτ. Και με τον κύριο Καντέκ βέβαια. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της σημαίας ευκαιρίας γιατί δημιουργεί προβλήματα κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γιατί είναι πολύ μικρά τα έσοδα των χωρών αυτών από τα πλοία μέση-μέση ευκαιρία. Για μεγάλες τέτοιες ε, χώρες μπορεί να φτάσει το ποσό των 10.000 ευρώ μόλις. Ακόμα και για μεγάλες χώρες που έχουν αλευτικά ε, ε, αλληλευτικά σκάφη μέση-μέση Ε, Και μάλιστα ε, χάνουν και τις ε, πρωτοπαραγωγικές τους πηγές, τα αποθέματά τους. Ε, οπότε ε, πλήττονται διπλά. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο αυτό το πρόβλημα για τον αναπτυσσόμενο χώρο από ότι για τον αναπτυγμένο πραγματικά. Συμφωνώ με την πρόταση της Ισαμπέλα για πιστοποιητικά που θα πιστοποιούν την νομιμότητα της αλίευσης των αλλιευμάτων και θα ακολουθούν τα αλλιεύματα σε όλη την αλυσίδα. Επίσης χρειάζονται ε, περιοδικές ε, αναθεωρήσεις της απόδοσης ε, των ε, ε, πόδα. Χρειάζεται επίσης διεθνή συνεργασία για να αποκτήσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και για τα αλλιευτικά σκάφη που ψάρεμουν σε διεθνή ύδατα και για τα σκάφη τα οποία κατηγορούνται για απλά. Και αυτές οι, αυτοί οι κατάλογοι θα πρέπει να αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται συνεχώς, όχι μόνο άπαξ ετησίως. Λοιπόν, είναι πολύ καλή αυτή βάση για, πολύ καλή βάση για την έκθεσή μας αυτή ε, η παρουσίαση. Κυρία Αντρές Μπαρέα. Θα συμφωνήσω με όλους και εγώ συγχαίρω την κυρία Λεβίν. Θα εξετάσω πολύ προσεκτικά αυτό το έγγραφο. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το κοιτάξουμε, είναι υποχρέωσή μας. Το πρόβλημα είναι ότι η νομοθεσία επιτρέπει τις σημαίες ευκαιρίας. Πρόκειται για θέμα διακυβέρνησης. Διακυβέρνησης με πολλούς τρόπους, Παγκόσμια διακυβέρνηση αλλά και διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, συγκεκριμένες καταστάσεις. Ε, συμφωνώ με την κυρία που λέει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το δικό μας το σπίτι. Αλλαγή της νομοθεσίας, να προσαρμόσουμε την νομοθεσία στην πραγματικότητα και ε, ενίσχυση, οικονομική ενίσχυση. Διότι χωρί ε, προπολογισμό δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μελέτες, ούτε να αποκτήσουμε στοιχεία, ούτε να συντηρούμε όργανα. Οπότε ε, αυτό ας το δούμε στην μελλοντική ε, μεταρρύθμιση της ελεκτικής πολιτικής. Οι ε, πόδα συνδέουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις άλλες χώρες και είναι σημαντικός ο ρόλος τους, θα πρέπει να τις ενισχύσουμε τις πόδα. Τώρα, σε σχέση με όσα είπε ο κ. Στίβενσον, ότι ο λιμένα στο Λασπάλμα, ε, ε, στην Ισπανία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί σημείο εισόδου παράνομη να του πω ότι αν έχει στοιχεία, παρακαλώ να τα βάλει στο τραπέζι. Μου το είπε μια φορά. Μου έστειλε και κάποια έγγραφα. Αλλά δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιγράφει ακριβώς. Είναι αλήθεια ότι εκφορτώνουν πλοία, αλλά είναι νόμιμη η εκφόρτωση. Δεν κάνουν τίποτα παράνομο. Οπότε επιτρέψτε μου ε, να αποφύγουμε την αμάυρωση ε, μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δεν σημαίνει τίποτα παράνομο εκεί. Γιατί εγώ πήγα στην Ισλανδία και παρόλο που μάλλον δεν παρανομεί, με εξέπληξε ε, η στάση της σε σχέση με τα εθνικά της συμφέροντα, χωρίς να κάνει τίποτα παράνομο. Και δεν ξέρω αν και στη Σκοτία συμβαίνουν πράγματα παράνομα ή όχι, τα οποία επιτρέπουν συγκεκριμένε οικονομικέ δραστηριότητε. Εγώ δεν έχω άλλε ερωτήσει, αλλά θα ρωτήσω κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά που διάβασα τι προάλλε τι δηλώσει τη κυρία Δαμανάκη στο Λονδίνο, λέγοντα ότι μπορεί να εγγυηθεί ότι όλε οι εισαγωγέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι λαθροαλία, πλά Έχω βέβαια τις αμφιβολίες μου ότι αυτό το οποίο είπε η κυρία Δαμανάκη θα ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Διότι... Αναφέρομαι εδώ στο έκτο κεφάλαιο για τις τρίτες χώρες, τις μη συνεργαζόμενες χώρες για την αναζήτηση μέτρων, για τη λήψη μέτρων σε μία, στα πλαίσια μίας τοπικής οργάνωσης αλίας κατά της ε, ΠΛΑ και εγώ το είπα και χθε όπου επέστρεψα από τον Ειρηνικό και όπου οι περισσότερες χώρες διαφωνούν και το αποδεικνύουν δηλαδή με τη συμπεριφορά τους, διαφωνούν ριζικά με την ε, λήψη οποιονδήποτε μέτρων ε, κατά της πλά. Ρωτώ λοιπόν αν αυτές οι χώρες οι οποίες δηλώνουν φανερά ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα και που έχουν αντιρρήσεις ε, να συνεργαστούν με τις τοπικές οργανώσεις αλίας ε, θα τους εφαρμοστεί το άρθρο 38 το οποίο απαγορεύει τις εισαγωγές διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως λέει και η κυρία Δαμανάκη ότι δεν εισάγει καθόλου προϊόν παράνομης αλίας και εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύετε ότι αυτό θα ισχύσει. Θα ήθελε και η Κομισιόν να συγχαρεί την εισηγήτρια. Η Κομισιόν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της έκθεσης και της προτάσεις. Πράγματι εσείς ε, τονίσατε ότι η καταπολέμηση της ΠΛΑ δεν θα έχει ε, αποτελέσματα άμα δεν, δεν καταπολεμηθεί διεθνώς πρόκειται για εγκληματική δραστηριότητα όπως το είπε και ο κύριος ε, Στίβενσον. Όπως είπε και ο κύριος Καντέκ πρέπει να πούμε ότι η μηδενική ανοχή θα πρέπει να εφαρμοστεί σε επίπεδο κοινοτική αγοράς και όταν τα διάφορα έγγραφα δεν συμπληρώνονται σύμφωνα με την νομοθεσία θα απαγορεύονται και εισαγωγές είχαμε περιπτώσεις ε, άρνησης απαγόρευση ε, απαγόρευσης συγγνώμη, εισαγωγών βάσει αυτού του συστήματος. Φυσικά τώρα κυρία Πρόεδρε η Κομισιόν εργάζεται για ελέγχους, για audit. Έχουμε ξεκινήσει διάφορους ελέγχους σε τρίτες χώρες για να επαληθεύσουμε την εφαρμογή του συστήματος των Kate Certificates σε αυτές τις χώρες. Και όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα προχωράμε σε διπλωματικά διαβήματα ούτως ώστε τα ε, ενδιαφερόμενα κράτη να αλλάξουν τακτική. Και όπως είπατε θα εφαρμόσουμε και το κεφάλαιο 6 και 5 του κανονισμού ΠΛΑ για να διαπιστώσουμε τις μη συνεργαζόμενες χώρες. Εμείς ερευνούμε ε, γύρω από πλοία με σημαία τρίτων χωρών αλλά και πλοία κοινοτικού ενδιαφέροντος και το πρόβλημα φυσικά είναι των δικών μας, των κοινοτικών που είναι μπλεγμένοι σε, αυτές τις, ε, σε αυτήν την αλή απλά. Εμείς θα εφαρμόσουμε την νομοθεσία κατά των εθνικών δηλαδή κατά των δικών μας παραβατών. Όπως επίσης θα κοιτάξουμε να βρούνε και τα ποια είναι τα πλοία με συμβατικές σημαίες. Οι τοπικές οργανώσεις αλίας προς στιγμή δεν έχουν αμέσα στη διάθεσή τους και εμείς θέλουμε να τις ενισχύσουμε ούτως ώστε να μπορέσουν να τιμωρήσουν τους συμβαλόμενους οι οποίοι δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό το οποίο θέλω να πω σε αυτή τη φάση είναι ότι θέλουμε να έχουμε μια εναρμονισμένη προσέγγιση τόσο μέσα και έξω από την Ένωση. Η κυρία Δαμανάκη δεσμεύθηκε για ανοχή μηδέν τόσο σε κοινοτικό επίπεδο χρήστες και πλοία όσο και τρίτες χώρες. Έχουμε ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόβλημα, ε, πρόγραμμα σήμερα και αυτό για τις επιθεωρήσεις και audit σε τρίτες χώρες και στις κοινοτικές χώρες. Και σας διασφαλίζω ότι εργαζόμαστε σκληρά γύρω από αυτό το θέμα και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Αλίας για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε που υπάρχει πρόβλημα και να εφαρμόσουμε τον κανονισμό πλά. Και βέβαια σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα του χρόνου να αναθεωρήσουμε όλη αυτή την νομοθεσία. Εμείς πάντως πιέζουμε τα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόσουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς και ούτω ώστε η μηδενική ανοχή να εφαρμοστεί στην Ένωση. Είναι πολύ σημαντική όλη αυτή η δουλειά. Βρισκόμαστε σε αναβρασμό. Όπως θα σας το πει και ο κύριος Κοστέρ σε λίγο, εμείς έχουμε ξεκινήσει ε, ε, διαδικασίες επιμόρφωσης στο Βίγκο ούτως ώστε να μπορέσουν να αφομοιώσουν όλους αυτούς τους κανόνες ή πλά είναι όργανο, γίνεται οργανωμένα. Πρέπει λοιπόν και η, να χρησιμοποιείται ο εφής έλεγχος και για να γίνει κάτι τέτοιο τα κράτη χρειάζονται κατάρτιση. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι το 2011 με αυτές τις νέες καταρτήσεις που δίνουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί κατά της ε, πλα αλίας και να εφαρμόσουμε τον κανονισμό και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και για τον κατάλογο των πλοίων που λαθροψαρεύουν αλλά και τις, να, να, επισημάνουμε και όλες τις δραστηριότητες λαθροαλίας. Να ενισχύσουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα σύμφωνα με την οδηγία. Ελπίζω να απάντησε. Κυρία Λόβιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Χαίρομαι που πολλοί και πολλές έθεσαν το θέμα των σημεών ευκαιρίας. Θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά και να βρούμε μια λύση. Είναι σκανδαλώδες. Φαινόμενο διεθνούς διάστασης. σημαίες ευκαιρίες και λιμές ευκαιρίες δεν είναι βέβαια φαινόμενο τόσο σημαντικό όσο η φορολογική παράδειση, αλλά θα πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστεί γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αυτό. Ε, ο κ. Καντέκ ρώτησε αν κυβερνήσεις δίνουν στατιστικά στοιχεία, ο καινούριο κανονισμός ε, ΠΛΑ ακριβώς αυτό έχει ως ε, στόχο, να μην μπαίνει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, την κατάλληλη, την επαρκή, τα, τα κατάλληλα έγγραφα. Μετά θα αξιολογήσουμε το κατά πόσον αυτά τα έγγραφα, τα συνοδευτικά έγγραφα, πραγματικά πιστοποιούν ότι το αλίευμα είναι νόμιμο. Και ε, αυτό είπε και η Κομισιόν ότι θα κάνει audit ελέγχου σε τρίτες χώρες για να διαπιστώσει το αν το σύστημα αυτό εφαρμόζεται και αν δίνει τα κατάλληλα αποτελέσματα. Χαίρομαι που ο κύριο Αρσένη συμφώνησε με την ιδέα για την ανεξάρτητο, ανεξάρτητο έλεγχο των ε, πόδα. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι βέβαια πολύ διαφανή για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και οι μαύρες λίστες θα, θα πρέπει να επικαιροποιούνται πολύ πιο συχνά. Κύριε Μπαρέα, Είναι σημαντικό να δούμε τι κάνουμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ εφαρμόζουμε τον κανονισμό πλά. Είναι βέβαια προφανές ότι όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια θα πρέπει να ενισχύσουν πάρα πολύ τις ε, ελεκτικέ τους ε, δραστηριότητες με μεγαλύτερους προπολογισμού, περισσότερου επιθεωρητές για να εφαρμόσουν σωστά τον κανονισμό πλά. Δεν μπορούν πλέον να δέχονται ε, έγγραφα χωρίς έλεγχο ή να επιθεωρούν μόνο το 10% των αλληλευτικών ε, σκαφών. Θα πρέπει ο κανονισμός να εφαρμοστεί ε, αξιόπιστα. Πώς είναι δυνατόν να ζητούμε από τους άλλους να φέρονται υπεύθυνα αν δεν φερόμαστε εμείς. Ευχαριστώ επίσης την Κομισιόν για τα σχόλιά της. Το επόμενο έγγραφο εργασίας ε, θα εξετάζει την διεθνή φυστάμενη νομοθεσία και τα παράθυρα, τα και τα οποία αφήνει. Θα εξετάζει τι πρόσθετα νομοθετικά κείμενα χρειαζόμαστε τι είδους νομοθεσία, για ποια θέματα, τι αδυναμίες προσπαθούμε να καλύψουμε. Βέβαια, είναι περίπλοκο, ε, όμως ε, ακολουθούμε μια σταδιακή προσέγγιση πριν την οριστική μας τελική έκθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόβιν θα υποβάλει μια, ένα δεύτερο έγγραφο εργασίας και μετά θα καθορίσουμε την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, μάλλον για τον Απρίλιο. Κλείνουμε και αυτό το θέμα. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Ε, Μαύρη θάλασσα. Ε, σημερινή και μελλοντική διαχείριση των ανακτικών δραστηριοτήτων στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ότοβα, κυρία Ιώτοβα, η συγγήτρια, είναι γνωμοδότη πρωτοβουλία μετά από αίτημα του, της ομάδας, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήδη έχετε το έγγραφο εργασία μου. Θα προσπάθησα στο έγγραφό μου να είμαι αναλυτική ε, για να μπορέσετε να δείτε διάφορες πτυχές ε, του θέματος της Μαύρης Θάλασσας. Είναι η πρώτη μας συνεδρίαση, η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και γι' αυτό ε, βασίζομαι στην άποψή σας για να είμαστε ακριβείς για τα διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με την αλία και την μαύρη θάλασσα. Κατανοείται ότι εύξηνος πόντος έχει ε, ως θέμα πολλές πτυχές. Δεν έχουμε ε, σκοπό να φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη στατιστική για τη λεκάνη, αλλά θέλουμε να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη της αλίας. Το 2011 θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και η έκθεση αυτή θα μπορέσει να συμβάλλει στην ολοκλήρωση του θέματος της ΚΑΠ λαμβάνοντας υπόψη ε, τις ειδικές ε, συνθήκες που επικρατούν στον εύξηνο πόντο, ο οποίος είναι εκτός της ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, ε, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Είναι ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2007 και σημαντικές πολιτικές αλλαγές που έγιναν μετά το 89 με την ε, κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και τα λοιπά ε, οδήγησαν στο να μην ληφθούν υπόψη ο εύξηνος πόντος και η περιοχή αυτή στην ΚΑΠ. Δεύτερον, ε, στον εύξηνο πόντο υπάρχουν δυναμικές αλλαγές στα οικοσυστήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της αλίας και την εξέλιξη της αλίας να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για έναν μία μη λεκάνη που έχει ε, μεγάλη περιοκτικότητα σε θιούχα και ανανεώνεται συχνά ε, με γλυκό νερό ε, Ε, και φυσικά ε, οι αληφτικοί πόροι ε, είναι, έχουν κατανεμηθεί μεταξύ των παράκτιων περιοχών, των κρατών εκεί. Στις πρώτες, στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 είχαμε μία μεγάλη πτώση της αλίας και μέχρι τώρα δεν μπορούμε να ανακάμψουμε αυτό διότι τα παραδοσιακά οικοσυστήματα, η μόλυνση και τα νέα ε, είδη όπως και η παραλίευση ε, ε, επιδίνωσαν την κατάσταση. Ο γάβρος, το σκουμπρί είναι είδη υποεξαφάνιση τα οποία μειώνονται σε απόθεμα συνεχώς ε, και οι προσπάθειες για αποκατάσταση δεν είχαν αποτελέσματα. Μειώνονται λοιπόν τα αποθέματα. Αυτό ισχύει για όλες τις χώρες που ακολουθούν τα ΤΑΚ, τα περιορισμένα ΤΑΚ, ε, με την εξαίρεση της Τουρκίας, η οποία δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο της αλίας της διαπραγματεύσεις της. Υπάρχει ένα πρόβλημα ε, με τις μη εγγεγραμμένες ε, μορφές ε, αλληλείας, ειδικότερα στην Ζωφική θάλασσα, είναι τεράστια τα ποσά. Γενικά ανέφερα τον τόνο, το σκουμπρί που αποτελούν πρόβλημα. Δεν έχουμε μία κοινή συμφωνία, έχουμε τη σύμβαση του Βουκουρεστίου και δεν έχουμε διμερείς ε, συμφωνίες που να είναι ξεκάθαρες. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία εφαρμόζουν την ΚΑΠ μετά το 2007 και το 2008 είχαμε ε, για το Καλκάνι και τον Ταούκι και, για, ε, και την Παπαλίνα για πρώτη φορά τα ΤΑΚ. Όμως οι υπόλοιπε χώρες δεν υποστηρίζουν αυτή την πολιτική ΤΑΚ και ποσοστώσεων και αυτό θέτει τη Βουλγαρία και την Ρουμανία σε πολύ διαφορετική θέση. Έχουμε παράνομο λοιπόν ανταγωνισμό και μη ε, ρυθμιζόμενες και καταγεγραμμένες, μη καταγεγραμμένες ε, αλλιεύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν την αναθεώρηση της ΚΑΠ και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής θα πρέπει να φτιάξουμε ε, τις κατάλληλες συνθήκες για να γίνει πιο ε, ακριβής ε, ερευνητική προσπάθεια για το οικοσυστήματα εκεί και την κατάσταση της θάλασσας. Έχω έρθω σε επαφή με εκπροσώπους από την ακαδημαϊκή κοινότητα και κανείς δεν έχει να μου δώσει σημαντικές πληροφορίες για το τι συμβαίνει στον εύξηνο πόντο. Χρειαζόμαστε λοιπόν άμεσα μέτρα για την απότομη μείωση των αποθεμάτων που είναι σημαντική όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά για όλη την περιοχή. Οι πόροι ε, μπορούν να βρεθούν στην επερχόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠΕ και το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2014. Η υποστήριξη λοιπόν της DG Mare και της ε, Επιτρόπου κυρίας Δαμανάκη ε, οι οποίοι προσπαθούν να έχουν συμφωνίες με κάποιες χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε τους μηχανισμούς για μια κοινή πολιτική μεταξύ των έξι χωρών που ε, βρέχονται από τον εύξηνο πόντο. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κοινή συμφωνία μεταξύ των χωρών αυτών ε, σημαίνει ότι ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ε, έγγραφο μια ανακοίνωση π.χ. της Κομισιόν που θα αγκαλιάζει τα συμφέροντα όλων των χωρών διαχείριση των αποθεμάτων, ε, κάτι που θέλουν οι δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Άγκυρα, όπως λένε οι συνάδελφοι από την Τουρκία. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει θεσμική δομή η οποία επαγγελματικά θα παρακολουθεί την αλία στον Εύξηνο Πόντο εδώ και δέκα χρόνια. Διαπραγματευόμαστε για τη μορφή και την εντολή μιας τέτοιας επιτροπής, για παράδειγμα, αλλά δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα ως τώρα και δεν υπάρχουν μέτρα για τον έλεγχο της αλληλείας και της ε, διασυνοριακής ε, αλληλείας. Η Γενική Επιτροπή για την Μεσόγειο δεν καλύπτει ε, αυτά τα στοιχεία υπάρχει αυτή η θέληση αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. μετά λοιπόν από διαβούλευση με την επιστημονική κοινότητα θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα δομή η οποία θα αντιμετωπίσει επαγγελματικά τα προβλήματα της ε, Μαύρης Θάλασσας. Να καταλήξω λέγοντας ότι η έκθεσή μου δεν θα συμβάλλει μόνο στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ αλλά και στην βελτίωση των σχέσεων με, τον, με τους ανατολικούς ε, ε, γείτονες. Ε, είχαμε το 2007 την ανακοίνωση της Κομισιόν για την συνεργασία στον Εύξηνο Πόντο που υπογραμμιζόταν η σημασία της αλίας και των τομεακών πολιτικών, ο συνάδελφος Κουρεάνο στο Στρασβούργο ε, κατέθεσε μια ε, έκθεση ε, την προηγούμενη εβδομάδα και η οποία έγινε αποδεκτή για, την, για τον εύξηνο πόντο και υπήρξαν κάποιες τροπολογίες στο έγγραφό του που υιοθετήθηκαν έτσι, σχετικά και η δική μου έκθεση θα μπορούσε να δώσει μια συστηματική αναθεώρηση για τις πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί που αναφέρονται σε διάφορα έγγραφα αλλά δεν είναι μέρος ενός γενικού συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ιώτοβα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Σε... Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με την ανάλυση που περιέχεται εκεί το πιο σημαντικό μήνυμα είναι νομίζω ότι ο εύξηνος πόντος ε, χρειάζεται μια συντονισμένη και περιφερειακή προσέγγιση στη διαχείριση της αλίας βασισμένη σε επιστημονική ανάλυση και στοιχεία. Από αυτή την έννοια δεν διαφέρει από άλλες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να τη μεταχειριστούμε διαφορετικά. Στην DG Mare έχουμε ξεκινήσει ε, τις εργασίες για μια περιφερειακή διαδικασία του Ευξήνου Πόντου, την ε, οποία θα συμπεριλάβουμε στην ε, ε, στρατηγική, στη συνολική στρατηγική της EAS. Νομίζω ότι χρειάζεται μια πραγματικά περιφερειακή στρατηγική για τον Ευξήνο Πόντο. Και μια τέτοιου είδους ε, στρατηγική θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη, ιδιαίτερο βάρος στην αλία. Ε, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ε, βάση για ένα καρποφόρο διάλογο με την Τουρκία, τη Ρωσία και με τις άλλες χώρες του Ευξήνου Πόντου. Η κυρία Δαμανάκη επισκέφθηκε και την Τουρκία και την Ρωσία και συζήτησε τον Ευξήνο Πόντο μεταξύ άλλων θεμάτων. Μάλιστα συμφωνήθηκε και με τις δύο χώρες να δοθεί συνέχεια στη συνεργασία. Ε, θεσπίζουμε ομάδες εργασίας και με την Ρωσία και με την Τουρκία λοιπόν αυτή τη στιγμή για να ε, δώσουμε συνέχεια σε αυτή τη συνεργασία, ιδιαίτερα στο θέμα της αλίας. Και εσείς ε, άλλωστε υπογραμμίζετε στο έγγραφό σας ότι ε, χρειάζονται, χρειαζόμαστε καλύτερες ε, επιστημονικές, καλύτερα επιστημονικά δεδομένα τα οποία θα βασίσουμε τις ε, αποφάσεις μας και δεύτερον, λέτε ότι χρειαζόμαστε ένα πιο διαρθρωμένο ε, πλαίσιο για την περιφερειακή διαχείριση της αλίας σε αυτή την ζώνη. Κάνετε και διάφορες προτάσεις μάλιστα ενδιαφέρουσες. Σε ό,τι φορά το πώς θα θεσπιστεί αυτή η περιφερειακή συνεργασία. Έχουμε ε, ε, αυτή η συνεργασία ε, έχουμε διάφορες αναλυτικές λύσεις, είτε την GFCM, ε, είτε μια ανεξάρτητη ε, οργάνωση. Η ε, GFCM της Μεσογείου δηλαδή περιλαμβάνει ήδη και την Γενική Επιτροπή Αλίας Μεσογείου, περιλαμβάνει ήδη και τη Μαύρη Θάλασσα, θα μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε ή να θεσπίσουμε κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό, ανεξάρτητο. Σε ό,τι φορά την επιστημονική βάση, Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ε, μακροπρόθεσμα, ένα ε, σύστημα το οποίο θα μας δίνει πληροφορίες ε, για τα αποθέματα καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα αλίας τακτικά και σίγουρα θα πρέπει σε αυτό το σύστημα να συμμετέχουν όλες οι παράκτιες χώρες του Ευξήνου Πόντου, οι παρευξήνιες χώρες. Έχουμε αυτή τη στιγμή επιστήμονες από την Τουρκία και την Ουκρανία που συνεισφέρουν ε, επιστημονικά και στην Επιστημονική Τεχνική Επιτροπή η οποία μας ε, συμβουλεύει ε, μαζί με τους, βέβαια, με τους εκπροσώπους της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση. σίγουρα χρειαζόμαστε μια συνεργασία έτσι ώστε να ε, συνδέσουμε μεταξύ τους τους διάφορους ε, ε, θαλάσσιους ε, τομείς, τομείς σχετικούς με την ε, θάλασσα. Ιδιαίτερα στην Μαύρη Θάλασσα χρειάζεται συντονισμός μεταξύ της IEP και της διαχείρισης αλληλείας. Θέλουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε με καινοτόμο τρόπο τους αλληλευτικούς πόρους έτσι ώστε να αυξήσουμε και την ανταγωνιστικότητα αλλά και να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση των παράκτητων περιοχών. Προσπαθούμε να βρούμε τους τρόπους αυτούς αυτή τη στιγμή. Όπως λέει η κυρία Ιώτοβα, η συνεργασία είναι η λέξη κλειδί προκειμένου να εξασφαλίσουμε ε, βιώσιμη διαχείριση των πόντων και σίγουρα θα συνεργαστούμε όλοι μαζί για να το πετύχουμε. Ε, η κυρία Ότοβα κάνει και συγκεκριμένε τεχνικέ προτάσει. Ε, πολύ ευχαρίστω θα τι ε, συζητήσουμε, αν το επιθυμείτε. Ιδιαίτερα στο, για το μακροχρόνιο σχέδιο διαχείριση. και εμεί υποστηρίζουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ μα ιδιαίτερος αν το επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σουκαλάς. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την κυρία Ιάτοβα για τη μέχρι τώρα συνεργασία και για τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που παρουσιάζει στο συγκεκριμένο άγγραφο εργασίας έχοντας λάβει υπόψη διάφορες απόψεις και οπτικές επί του θέματος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εστιάσω κυρίως σε ορισμένα θέματα, τα οποία θεωρώ ιδιαίτερο σημαντικά. Καταρχάς, όπως αναφέρει και η συγγήτρια, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης της επιστημονικής έρευνας, ούτως ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται και έχουν άμεσες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαντολογικές συνέπειες να βασίζονται σε τεκμηριωμένα και βάσιμα στοιχεία. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ιδιαίτερο το γεγονός ότι όλα τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας και κυρίως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υποψήφια για ένταξη κράτη οφείλουν να σέβονται τη σχετική κοινοτική νομοθεσία κατά την άσκηση των αλλιευτικών και μη δραστηριοτήτων και να στοχεύουν στη βιωσιμότητα όχι μόνο των αλλιευτικών αποθεμάτων αλλά και του αλλιευτικού τομέα. Σε αυτό θα μπορούσε να προσθεθεί και ο σημαντικός ρόλος των διμερών συνεργασιών και των διεθνών συμφωνιών, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με τη δημιουργία ξεχωριστού φορέα για τη διαχείριση της αλίας στον αύξηνο Πόντο, θεωρώ ότι πρόκειται για μια αξιόλογη αλλά αρκετά φιλόδοξη ιδέα. Όντως υπάρχει ανάγκη, όπως αναφέρει και η αξιότιμο συνάδελφος, να βρει ο εύξηνος πόντος τη θέση που του αξίζει στην κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεω και η εν λόγω λεκάνη να αντιμετωπίζεται επί ίσης όρις με τις άλλες λεκάνες. Παρόλα αυτά, η δημιουργία ενός ξεχωριστού φορέα ίσως δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Μια εναλλακτική λύση θα μπορούσε ίσως να είναι μια εξειδικευμένη ομάδα εργασίας εντός του πλαισίου της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, στην οποία θα συμμετείχαν εκπρόσωποι και από τα έξι κράτη-μέλη της Μαύρης Θάλασσας. Σχετικά με την πρόταση κατάργησης της υφιστάμενης αρχής ετησίων συνολικών επιτροπομένων αλλιευμάτων και ποσοστώσεων, που έχει επιβληθεί στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και την αντικατάστασή του από ένα πολιετές σχέδιο διαχείρισης Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα, αλλά φοβούμε ότι δεν θα γίνει εύκολα δεκτή η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, σχετικά με το θέμα της αλληλεία με τράτα, θα συμφωνήσω με την εισηγήτρια πως για να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση υπέρ ή κατά της κατάργησης της χρήσης της, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επιστημονικές έρευνες και οι ενδεχόμενες συνέπειες για την οικολογική κατάσταση του ευξήνου πόντου και την ευημερία των αλλιέων στη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ομολογουμένως χαρακτηρίζεται από ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες. Αυτές τις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Τα παραπάνω σχόλια παραμένουν βέβαια πρώτες σκέψεις σχετικά με τη διαχείριση της αλίας στη Μαύρη Θάλασσα και δεν χρειάζεται πιστεύω να αναφέρω ότι παραμένω πρόθυμος και ανοιχτός για κάθε συζήτηση. Σας ευχαριστώ. para η κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Έχουμε καλή συνεργασία. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ε, απαρχή δημιουργίας μιας νέας πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κοινότητα. Οι στόχοι που θέσαμε ε, οι ίδιοι μπορεί να φαίνονται εξ αρχής κάπως φιλόδοξοι. Όμως ε, σας διαβεβαιώ ότι πρόκειται για ένα καλό πρώτο βήμα. Αυτή τη στιγμή από τη συζήτηση που έγινε γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια νέα πολιτική για την ε, ανάπτυξη της πολιτικής. Η εξέλιξη της αλίας και ανάπτυξη της αλίας είναι ε, ε, μια καλή εξέλιξη για την περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους από την Επιτροπή Αλίας που με υποστήριξαν στην έκθεσή μου και για όσους ενδιαφέρθηκαν θεωρώ ότι μπορούμε να συμβάλλουμε. Ωραία. Θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα στις 15 και 16 Μαρτίου. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έκθεση The Gallagher. Απαλλαγή 2009, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ελέγχου Αλληλείας του Βίγο. Ξέρω ότι δεν είναι παρόν. Δεν είναι παρόν ο κ. Γκάλαγκερ. Χρειάστηκε να γυρίσει στην ε, χώρα του πηγόντος. Είναι πολύ απλή η γνωμοδότηση, ε, η έκθεσή του επιβεβαιώνει κατά βάση ότι το ελεκτικό συνέδριο ε, υπογράμμισε πως ο προϋπολογισμός 10 ε, ευρώ απεικονίζει ε, πιστά, μάλλον ο λογαριασμό για τον προϋπολογισμό απεικονίζει πιστά τα αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του χαρακτήρισε νόμιμες και κανονικές οικονομικές καταστάσεις υπηρεσίας για το έτος 2009 και εγκρίνει την απαλλαγή. Δεν δημιουργεί κανένα θέμα αυτή η γνωμοδότηση. Προθεσμία για τροπολογίες λοιπόν 4 Φεβρουαρίου. Θα ψηφιστεί στην Επιτροπή στην συνεδρία στις 15 Μαρτίου. Το σημείο 15 έχει αναβληθεί η απόφαση που λάβαμε χτε. Στα διάφορα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, αν όχι να περάσω στο σημείο 17, ανακοινώσει της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές. Θα σας αποσταλούν από την γραμματεία αμέσω μετά τη συνεδρίασή μας και θα τις ψηφίσουμε, θα τι εγκρίνουμε την επόμενη εβδομάδα. Τέλος. Σημείο 18, ημερομηνία τη προσεχού συνεδριάσεως, 1η Φεβρουαρίου 2011, 9 με 12 και 3 με 6.30 το απόγευμα, στις Βρυξέλλες. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Και κύριε ότι συνεδρίασης.